Αγαπητοί συνάδελφοι, να μην τιμωρήσουμε αυτούς που ήρθαν στην ώρα τους, οπότε να ξεκινήσουμε. Δευτέρα απόγευμα στο Στρασβούργο, το γνωρίζω. Είναι κάπως δύσκολο. Αλλά οι ενδιαφερόμενοι, πραγματικά ενδιαφερόμενοι είναι εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν με το σημείο της μερισιάς διάταξης, έγκριση δηλαδή του σχέδιου μερισιάς διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσει ό,τι αφορά τη μερίσια διάταξη. Όχι, επομένω εγκρίνεται η μερίσια διάταξη ό,τι αφορά τι ανακοινώσει τη Προέδρου. Θέλω να σα πω τα συνήθη, Καταρχά δηλαδή ότι έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας διερμηνία στι εξή γλώσσε. γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσέχικα, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά και ρουμανικά και να σα πενθυμίσω επίση όπω πάντα ότι η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Περνάμε τώρα στο σημείο 3 της μερίσιας διάταξης. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον κύριο Σάντζιους. Αφιβάλλω να το πρόφερα σωστά το όνομά σα και λυπούμε γι' αυτό. Καλωσορίζω πάντω τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ελληνικτικού Συνεδρίου, που είναι συντάκτη τη ειδική έκθεση του Συνεδρίου για το Erasmus Plus έκθεση η οποία αναλύει το πώς έχει εφαρμοστεί το τρέχον πρόγραμμα Erasmus Plus και θα μας δώσει φαντάζομαι και ο συγητής ε, σημαντικά στοιχεία για την διαμόρφωση του νέου, τη νέα πρόταση για το νέο Erasmus. Έχουμε επίσης βέβαια και τη δική μας έκθεση που ακολουθεί θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάτζιους ή κάπως έτσι. Έχετε λίγο πολύ 10 λεπτά στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ιδιαίτερη τιμή για εμένα να είμαι εδώ. Αλλά δεν μιλάω τόσο καλά γερμανικά. Οπότε αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω αγγλικά. Κανένα πρόβλημα λέει πρόεδρος αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι συνάδελφοι από τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα, νομίζω ότι είναι εύκολο το σημερινό μου έργο, διότι έχουμε δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη αυτή τη συνεδρίαση ε, από κοινού. Το ένα είναι η δική μας ειδική έκθεση και νομίζω ότι ε, ταιριάζει πολύ καλά με το επόμενο θέμα της μερισιάς διάταξης, την έκθεση για τη νέα νομοθεσία για το Erasmus ή Erasmus Plus, Erasmus Sin, όπως πρότεινε ο εισηγητής. Πολύ γρήγορα λοιπόν να σας ε, περιγράψω κάποιες ε, διαφάνειες που ενδεχομένως σας προκαλέσουν απορίες, με τα χαράς να απαντήσω στη συνέχεια το Erasmus. Λοιπόν, εμείς μελετήσαμε και κάναμε τον ε, λογιστικό έλεγχο μόνο για το ένα, την ε, πρώτη δράση του Εράσμους και τα επόμενα λεπτά μόνο για αυτή τη δράση θα σας μιλήσω, δηλαδή την ε, μαθησιακή κινητικότητα, το Learning Mobility. Είναι ένα πρόγραμμα που συνδυάζει πολλές δράσεις και 33 χώρες ε, με διάφορες δομές, διάφορα φορείς, 28 ε, τα μέλη της Ένωσης, συν 5, 145 χώρες εταίρους επίσης. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά τα νούμερα, ουσιαστικά καλύπτουμε... It is indirect management ε, which makes some problems in spending. Πρόκειται για άμεση διαχείριση, οπότε υπάρχουν κάποια προβλήματα. our aim was... Ο στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε την αξιολόγηση και την προσθέμενη αξία του προγράμματος. Γιατί? Διότι ήταν δύσκολο εμείς να ελέγξουμε ένα θετικό πρόγραμμα που όλοι δηλαδή το αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά ε, στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να βασιστούμε στα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο. Και εμείς αυτό που θέλουμε είναι να δούμε ακριβώς λεπτομεριακά τι θα πει ακριβώς ε, προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία που είναι μια κοινοτοπία για τους ε, πολιτικούς όμως ε, δεν είναι και πάντοτε ακριβώς αντιληπτό τι σημαίνει. Το δεύτερο ήταν η επιδόσεις, η απόδοση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για να δούμε πώς δουλεύει το πρόγραμμα γιατί στο μέλλον, στο μέλλον προβλέπεται αυξημένη χρηματοδότηση. Τι διαπιστώσαμε, ότι είναι ένα καλό, επιτυχημένο εμπορικό σήμα. Και το τονίζω αυτό. Έγινε εμπορικό σήμα, ε, σήμα σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μια μάρκα. Ήταν ε, το ευρώ που το συναγωνιζόταν, αλλά τώρα είναι πιο γνωστό αυτό το, αυτό το εμπορικό σήμα. Πρέπει όμως να το προωθήσουμε κιόλας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έτσι τα πράγματα και πρέπει να το... Νομίζω δεν υπάρχει μετάφραση στα Ιταλικά. No? Also, French is not... Δεν δουλεύουν οι μεταφράσεις. Πράγματι έκλεισε το μικρόφωνο όλων των καμπινών πριν από λίγο. Français, okay? Okay try another uh headphone okay vielleicht können die να πούν κάτι οι Ιταλοί συνάδελφοι για να βεβαιωθούμε ότι ακούγεται η Ιταλική δερμηνία. Ωραία. Εντάξει, όλα πάνε καλά τώρα. Ωραία, άρα μπορώ να συνεχίσω. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να δούμε πώς το πρόγραμμα αυτό ε, το Erasmus Plus παράγει προσθέμενη αξία. Και κάνοντας αυτή την ε, μελέτη βρήκαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχουν αυτά που περιγράφει ο κανονισμός, ε, αλλά υπάρχει προσθέμενη αξία που ξεπερνά πολύ τις νομικές απαιτήσεις. Θα σας δώσω παραδείγματα που αποκονίζουν αυτό που σας είπα. Η διασυνοριακή προσέγγιση, ε, και άλλα. Τα λέει ήδη το πρόγραμμα. Εντάχθηκε όμως και στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Η ήπια διπλωματία. 145 χώρες. Γι' αυτό δόθηκαν από τους συνομοθέτες από τη γραμμή των εξωτερικών δράσεων κάποια κονδύλια παραπάνω. Λογικό αυτό. Όμως όταν σκεφτόμαστε χρηματοδότηση των προγραμμάτων ε, των μελλοντικών στο πλαίσιο του Erasmus Plus, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το έξτρα αυτό αποτέλεσμα. Κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον. Είναι οι χάρτες των ευρωπαϊκών ε, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στην περίπτωση των ιδρυμάτων ανώτερης ανώτατης εκπαίδευσης, Υπάρχουν κάποιοι φορείς που δεν θέλουν να συμμετέχουν ε, στο Erasmus Plus, αλλά ε, κάνουν έτσι για το χάρτη γιατί θεωρούν ότι είναι ε, από ποιοτική πλευράς κάτι απαραίτητο. Και αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο. Και ένα άλλο υποπροϊνόρνα, η παράγωγο προϊόν, παράγωγη αξία που βρήκαμε είναι αυτό το σχήμα που σας περιγράφω. Τεράστια αύξηση της ε, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σπουδαστών δηλαδή που συμμετέχουν από την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση στο Erasmus Plus, ακόμα και σε αυτή την περίοδο δηλαδή. Προσέλκυσε σπουδαστές που δεν είναι τόσο ε, επιτυχημένο το υπόβαθρο από το οποίο προέρχονται ή τέλο πάντων δεν αποσκοπούν στο να αποκτήσουν κάποιο δίπλωμα ανώτετα της εκπαίδευσης. Θέλαμε λοιπόν να δούμε τι προτεραιότητες ε, θα ε, είχαμε να ε, προτείνουμε. μεταξύ άλλων και για τη χρηματοδότηση. Μέτρηση της επίδοσης, της απόδοσης. Ειδική και γενική είναι η στόχη. Ποιοι είναι οι γενικοί στόχοι καταρχάς και για τους ε, σπουδαστές και για το προσωπικό. Πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες, να αποκτήσουν εργασιακή πείρα στο εξωτερικό. Για τους διάφορους φορείς, ποιότητα, καινοτομία, αριστεία, διεθνοποίηση. Υπάρχουν όμως και ειδικοί στόχοι. Η μαθησιακή κινητικότητα είναι αυτό το οποίο εγώ θα τόνιζα ιδιαίτερα. Ελέγξαμε και είδαμε ε, ότι υπάρχει και ο κίνδυνος να γίνει απλά τουρισμός η μασική αυτή κινητικότητα, η κινητικότητα των σπουδαστών. Όμως στην πράξη δεν αποκρισταλώνεται έτσι. Τις περισσότερες φορές τα μόρια που παίρνουν ε, δουλεύει το σύστημα το εξωτερικό. Υπάρχουν κάποια παράπονα. Θέλουν ε, οι σπουδαστές να περάσουν καλά εκεί που πάνε. Ε, τέλο πάντων, με θεσική κινητικότητα είναι κάτι ενδιαφέρον. Επίση, για τη μέτρηση των επιδόσεων, τι θα τόνιζα εγώ. Αν έχουμε ένα πρόβλημα, ή γιατί τέλο πάντων έχουμε θέσει κάποιου στόχου, η απάντηση των πολιτικών πάντα είναι χρήματα. Να δοθούν χρήματα. Έχουμε κάτι μεταξύ όμως των στόχων και του χρήματος. Αυτά είναι βαρετά ίσως οι δείκτες, μέτρηση δηλαδή των επιδόσεων, κάποιοι μηχανισμοί. Ούτε η πολιτική ούτε και το πλάτη κοινό φαίνεται να δείχνει τόσο ενδιαφέρον για αυτά. Αλλά χωρί αυτά δεν θα λειτουργούσε το σύστημα. Είδαμε λοιπόν ότι πράγματι περισσότεροι στόχοι που ετέθησαν για τους δείκτες ε, εκπληρώνονται. Δεν είναι όμως κατάλληλοι για να μετρήσουν το συνολικό αντίκτυπο, την έκβαση, το αποτέλεσμα των προγραμμάτων επηρεάζουν την απασχολησιμότητα, την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, ε, την ολοκλήρωση του ε, συστήματος ε, του εκπαιδευτικού των κρατών μελών. Άρα πρέπει να βελτιωθεί αυτό το στοιχείο και να δοθεί τεράστια προσοχή σε αυτά τα έστω βαρετά, πολύπλοκα θέματα. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν έχουν δεξιότητες πάλι της Κομισιόν, απλά είναι πολύπλοκο το θέμα. Αξίζει όμως να το μελετήσουμε και χαίρομαι που στην έκθεση που θα συζητήσετε εν συνεχεία ήδη προβλέπονται κάποια μέτρα, κάποια βήματα για το σκοπό αυτό. Απλούστευση καινοτομία. Πολλά ζητήματα μελετήσαμε. Είδαμε ότι υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις ε, σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα σε αρκετά σημεία. Απλούστευση υπάρχει λοιπόν η διαδικασία όμως πώληση αιτήσεων ε, και αξιολόγηση εξακολουθεί να παραμένει πολύπλοκη. Πολύ φορτωμένη ενίοτε με αυτή την ευρωπαϊκή τεχνική ορολογία, την αργό που ούτε μπορούν ούτε και θα έπρεπε να μπορούν να καταλαβαίνουν οι σπουδαστές από την αρχή. Άρα προτείνουμε να υπάρξει μια περαιτέρω απλούστευση. Η υποβολή αναφορών ενίοτε βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση. Δεν μπορούμε να το καταλήψουμε αυτό, πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Όμω, θα πρέπει να αξιολογήσουμε σωστά και τα αποτελέσματα. Η διδασκαλία σε αίθουσα διδασκαλία ε, είναι και αυτό κάτι πρέπει να προτείνουμε. Πολλέ φορέ, α πούμε, γλωσσικέ δεξιότητε ελέγχονται με ένα σύστημα online. Πριν ξεκινήσει το Erasmus, η διαμόνη στο εξωτερικό. Και κάποιε φορέ δεν είναι καλά τα αποτελέσματα. Ε, είναι διαφορετικά τέλος πάντων. Κάποιοι το βλέπουν ως μία διατύπωση, ως κάτι τυπικό, αλλά νομίζω ότι με την αίθουσα και το μάθημα σε αίθουσα ε, μπορεί πραγματικά ο σπουδαστής να αποκομίσει μια αίσθηση της πολυγλωσσίας κτλ. Ε, θέλουμε και οι διδακτορικοί φοιτητέ να συμμετέχουν και αυτό δεν είναι απλό, γιατί το διδακτορικό παίρνει χρόνο. υπάρχουν προβλήματα πολλές φορές. Και κάτι άλλο το οποίο συνιστούμε είναι και οι μαθητές των σχολείων να περιληφθούν στο πρόγραμμα κινητικότητα του Erasmus+. Και θέλω να ευχαριστήσουμε την Κόμιση που ακόμα και πριν δημοσιοποιηθεί έκθεση εισήγαγαν αυτό το σημαντικό στοιχείο στο πρόγραμμα. Και με αυτό το ευχάριστο, με αυτήν την ευχάριστη νότα ολοκληρώνω την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την γρήγορη αυτή επισκόπηση των αποτελεσμάτων και ήδη νομίζω με την πρώτη ματιά βλέπουμε ότι πολλά ε, από αυτά που περιλαμβάνει η έκθεση είναι αυτά τα οποία μας βρίσκουν σύμφωνος, τα έχουμε συζητήσει ε, και από το feedback που παίρνουμε. Δηλαδή ότι πράγματι ε, είναι καλό και έχουμε και την ε, επιβεβαίωση τώρα από το ελεγκτικό συνέδριο. Και σε ό,τι αφορά τα προβλήματα τα οποία έχουμε και εμείς επισημάνει ή μας έχουν μεταφέρει. Νομίζω ότι και αυτά ακριβώς ε, τα έχει ίδια, τα ίδια ακριβώς πρέπει να τα έχει επισημάνει και το ελεγκτικό συνέδριο. Και υπάρχουν και κάποιες συστάσεις και προτάσεις ε, για το νέο πρόγραμμα, για να υπάρξουν ακόμη περισσότερες βελτιώσεις ή ε, απλούστευση, ε, όχι μόνο των αιτήσεων, γιατί αυτό είναι κάτι πολύπλοκο, είναι σε μια γλώσσα που οι νέοι ίσως δεν την καταλαβαίνουν και όλα όσα είπατε για την υποβολή αναφορών και είναι ενδιαφέρον να το λέει και το ελεγκτικό συνέδριο ε, και επίσης τι γίνεται με τα χρήματα, κατά πόσον πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Και λέτε κι εσείς επίσης ότι θα μπορούσε να αποπλουστευτεί ακόμη περισσότερο η υποβολή των αναφορών. πρέπει να αποδειχθεί ότι τα χρήματα έχουν ταπανηθεί σωστά το Ελληνικό μισθό. τα λέει και η ε, δική σας πλευρά τα ίδια, ε, το Ελληνικό Συνέδριο ζητάει και εδώ απλούστευση, είναι καλό το αποτέλεσμα για μας. Θα ήθελα τώρα, εντάξει δεν είμαστε και τόσοι πολλοί, όχι τόσο επίσημα, Στα θα μπορούσαμε και τυπικά να συζητήσουμε, αλλά ε, δεν είμαστε πολύ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για το Εράσμου, στον κύριο Σβέρ και από εκεί πέρα όποιος άλλος θέλει να κανει παρατηρησει παρατηρήσεις. Κύριε Σβέρ, δύο-τρία λεπτά και θα έχετε πιο πολύ χρόνο μετά όταν έρθει το σημείο που θα συζητήσουμε τη δική σας έκθεση. Ε, Ευχαριστώ για το λόγο. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Λεκτικού Συνεδρίου για την εξαιρετική παρουσίαση. Είναι μεγάλη η τιμή μου. Μόλι πριν λίγες εβδομάδες είχα μια εξαιρετική συζήτηση μαζί του. Έμαθα πάρα πολλά για την ευρωπαϊκή έννοια της ευρωπαϊκής προστατεμένης αξίας ε, και είναι πολύ μεγάλη τιμή να μαθαίνω από τη δική σας σοφία. Εγώ πιστεύω ότι το Erasmus Plus και οι διεθνείς ανταλλαγές ε, έχουν ε, πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτά που μπορούν να δείξουν οι στατιστικές ή οι, οι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορείς να τα αναλύσεις όλα με νούμερα ή με στατιστικά στοιχεία η προσθέμενη αξία σε ό,τι αφορά το Erasmus Plus είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης ε, όψεως με αριθμητικά στοιχεία. Ε, ευχαριστώ πολύ το Ελεκτικό Συνέδριο για την έκθεσή του, κυρίως ε, για τις συστάσεις ό,τι αφορά την απλούστευση. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να μειώσουμε το διοικητικό άχθος και αυτό είναι ένα μέρος του Erasmus όλο αυτό το άχθος έχει καταστήσει πάρα πολύ δύσκολη τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους. Ακόμη και αν ε, μιλάμε για ένα πρόγραμμα μικρής διάρκειας, θα πρέπει να επενδύσεις πάρα πολλά σε διοικητικό επίπεδο και φυσικά αυτό αποτελεί εμπόδιο και είμαι σίγουρος ότι θα εξεύρουμε μια καλή λύση με τη συνεργασία με το Λεκτικό Συνέδριο. Σίλβια Κώστα. Σας ευχαριστώ, Σίλβια Κώστα. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σα. Ζητώ συγγνώμη γιατί η συνάδελφο Λιγκά Μπάτσκα, που είναι η συγγήτρια και τη οποία θα διαβάσω την έκθεση, οικογενειακού λόγου δεν μπόρεσε να παραστεί. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα δύο-τρία σημεία. Πρώτον, λέτε ότι ευτυχώς παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση κατά 34% της επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό επανέφερε μια ισορροπία και είναι πολύ σημαντικό. Λέτε και κάτι άλλο που με βρίσκει σύμφωνη, ότι θα πρέπει να δώσουμε στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μεγαλύτερο περιεχόμενο. Μιλάμε για την ευρωπαϊκή κατάρτιση, αλλά για πιο ε, ε, τυποποιημένη συμμετοχή σε επίθετο γλώσσα. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι αυτό έχει συρρυγνωθεί. Τρίτη ερώτηση. Αναφερθήκατε στο θέμα των ανθρώπων που προέρχονται από ένα προβληματικό πλαίσιο. Ζητήσατε να υπάρχει μια μεγαλύτερη εναρμόνιση των κριτηρίων γιατί κάθε χώρα ερμηνεύει διαφορετικά με την έννοια του προβληματικού. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα άτομα και πώς θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τα δεδομένα. Η συνάδελφος Λιμπάσκα θεωρεί ότι η πρόσβαση σε αυτά τα άτομα είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Τελευταίο σημείο. Λέτε ότι όντως δεν πήγε καλά η ευρωπαϊκή εγγύηση για το δάνειο στους φοιτητές. Εσείς ως ελεκτικό συνέδριο θα είχατε κάποια πρόταση να κάνετε, έχετε κάτι να μας πείτε για το πώς τάσαμε σε αυτό το σημείο. Julie Ward, Julie Ward. Ah, thank you very much uh, Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Εν μέρη βρίσκομαι εδώ γιατί ήμουν ε, φοιτήτρια στο Erasmus Πράς και συνεργάστηκα και με περιθωριακές κοινότητες. Η δική μου εμπειρία φορούσε άτομα που ήταν εκτός ενός κοινωνικού πλαισίου. Ε, άτομα που διέτρεχαν κίνδυνο να έχουν προβλήματα με το νόμο, που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την ένταξη στην κοινωνία και στην κοινότητά τους. Εγώ συνεργάζομαι με μία παλιά ε, κοινότητα ανθρακορίχων και δεν έχει ε, εμπειρία επαφής με άτομα από άλλες χώρες. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία και αυτό έγινε στα πλαίσια ενός προγράμματος δράσης πριν καν αποκτήσει το όνομα Εράσμους. Η δική μου άποψη είναι τις ε, ζωές αυτών των ανθρώπων, τις μεταμόρφωσε η επαφή με άλλους νέους. Απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ακόμα και μετά τη συμμετοχή δεκαπενθύμερου προγράμματος ε, στη Γερμανία. Τα παιδιά αυτά απομακρύθηκαν από την, τον τόπο τους, μεταμορφώθηκαν, ε, απέκτησαν δουλειές, ασχολήθηκαν με τον εθελοντισμό, ασχολήθηκα με την εκπαίδευση και είναι σημαντικό γιατί τους ανθρώπους αυτούς τους παρακολουθώ, έχω επαφή μαζί τους 10-15 χρόνια μετά. Μιλάω λοιπόν για κάτι απόλυτα αυτό. Μετά την εκλογή μου είχα το προνόμιο να σταθώ μάρτυρας της εφαρμογής μιας σειράς προγραμμάτων με τα παιδιά αυτά. Θα ήθελα να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Νέα άτομα που πάσχουν από αυτισμό. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν εύκολα να ε, συνεννοηθούν με τους συνομιλίκους τους, δεν αρέσκονται σε νέες εμπειρίες και υπάρχει στη δική μου περιφέρεια ένα σχολείο ε, τα παιδιά μου αυτά δεν τα συνάντησα στο Μάντσεστερ, τα συνάντησα στις Βρυξέλλες, γιατί πήραν μέρος στο πρόγραμμα εράσμους και μετά τα συνάντησα και στο σχολείο του στο Μάντσεστερ. Τα παιδιά αυτά είχαν αποκτήσει και εκεί πήρα ήξεραν να γράφουν τα βιογραφικά τους, έστησαν επιχειρήσεις. Ήθελα λοιπόν να σας τα πω αυτά, γιατί πολύ συχνά όταν αναφερόμαστε στο Erasmus πλάσα δίνεται ε, η εντύπωση ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν αυτοπεποίθηση και πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρουν όμως για την ύπαρξη άλλων προγραμμάτων. Αυτά τα προγράμματα υπάρχουν και υπάρχουν και άτομα που δρούν ως πρεσβευτές, ε, πρεσβευτές του προγράμματος και πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταβάλουμε μια προσπάθεια να έχουμε στα χέρια μας όλα αυτά τα δεδομένα, τα στοιχεία για να μιλήσουμε στους ανθρώπους. Δεν είναι ένα πρόβλημα, ένα πρόγραμμα που αφορά τους λαμπερούς που σε κάθε περίπτωση θα πήγαιναν στο πανεπιστήμιο. Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται και σε περιθωριοποιημένα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν δεδομένα για να μπορέσουμε να δείξουμε πόσο επιτυχές ήταν αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση από δική μου πλευράς. Μιλήσατε για τους δίκτες με τους οποίους μετράμε την επιτυχία. Ότι θα πρέπει να τους φέρουμε λίγο πολύ σε ε, ευθυγράμμιση με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, γιατί ακόμα δεν είναι τόσο καλή. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν να είναι πιο ακριβείς ε, και αποτελεσματικοί δείκτες. Ε, έχετε ιδέες και έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω την αίσθηση ότι παρουσίασα ένα πρόγραμμα για το μέλλον των καθήκων, όμως ε, των μελών του ελεκτικού συνεδρίου είναι διαφορετικό. Οι ελεκτέ είναι μάλλον δυσάρεστα άτομα που παραθέτουν γεγονέτοντα και μετά ε, κάνουν ε, γενικές συστάσεις και μία από αυτές τις συστάσεις απευθυνόταν στην Επιτροπή και αφορούσε το σύστημα των δικτών. Η γενική θεωρία λέει ότι υπάρχουν εισερχόμενα δραστηριότητες, εξερχόμενα που ελέγχονται εύκολα. Αλλά είναι δύσκολο να μετρηθεί το αποτέλεσμα και το, τα έσοδα από ένα πρόγραμμα. Ήδη καταβάλλονται μερικές προσπάθειες στην Επιτροπή προκειμένου να καταλάβουν τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την, ε, το ποσοστό απασχόλησης αυτών των ατόμων, ε, δηλαδή βελτιώνεται η, απασχολησιμότητά τους. Ε, έχουν φτιάξει μια βάση δεδομένων των αποφοιτησάντων και τους παρακολουθούν κατά την διάρκεια της ζωής τους. Η κυρία Γουότς παρέθεσε ένα παράδειγμα και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να συγκρίνουμε με άλλους φοιτητές που έχουν ένα παρεμφερές, μια παρεμφερή καταγωγή, ένα παρεμφερές υπόβαθρο. Βεβαίως, αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Θα πρέπει κανείς ε, να περιμένει για να δει τι συμβαίνει. Ε, κάποιοι άλλοι ε, με ρώτησαν αν το Erasmus Plus είναι σχεδιασμένο προκειμένου να προωθήσει την απασχολησιμότητα των νέων στο εξωτερικό. Επουδενή όχι. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι η απασχολησιμότητα των νέων, η δυνατότητα να βρουν μια καλύτερη δουλειά στο σπίτι τους και όχι σε μια ξένη χώρα. Αλλά βεβαίως ε, η μελέτη των αποφοιτησάντων θα είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως είπε η κυρία Τώρα, ένα άλλο θέμα αφορά τα άτομα που προέρχονται από ένα προβληματικό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που συναντάται σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής, ε, της, του κόσμου, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαστρωμάτωση της κοινωνίας αναπαραγάγεται στα ανώτατα εκπαιδευτικά συστήματα. Πώς είναι δυνατόν να αναμειχθούν όλοι αυτοί οι νέοι. Πιστεύω ότι το Erasmus Plus απευθύνεται σε νέους που είναι στο σχολείο ή που παρακολουθούν μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, άτομα δηλαδή που δεν έχουν μια ξεκάθαρη κοινωνική θέση. Και η, και η παρέμβαση του Εράσμου σε αυτή τη φάση νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Τώρα, ε, ε, κάτι άλλο που παρατηρήσαμε ε, εμείς και ο εισηγητής ο κύριος ε, Σβέλ για την ε, μελλοντική νομοθεσία. Η παράγραφος 66 της έκθεσής μας αναφέρει ο ορισμός των ε, μειονεκτούντων ατρόμων διαφέρει σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, στην Ισπανία τα άτομα που παίρνουν επίδοση, επίδομα για τις σπουδέ συμπεριλαμβάνονται εδώ. Τα δεδομένα λοιπόν από τις διάφορες χώρες δεν είναι συγκρίσιμα. Όταν παρουσίασα αυτή την έκθεση στο Συμβούλιο, ε, στην Επιτροπή ε, Παιδείας, διαπίστωσα ότι ότι δεν θέλουν, ε, δεν είναι πρόθυμες ε, οι διάφορες χώρες να επιτευχθεί μία εναρμόνιση σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες. Πιστεύω όμως ότι μία στο εν εναρμόνιση με κατεξουσιοδότηση νομοθεσία ή συμπεριλαμβάνοντας όπως πρότεινε ο κύριος Βερ τουλάχιστον μερικά κριτήρια, μερικές ενδείξεις στον κανονισμό θα μπορούσε να ε, βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όλες ε, ε, οι χώρες θέλουν να τα εκπαιδευτικά τους συστήματα να λειτουργούν καλά και με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται μία άμυλα, ένας ε, ανταγωνισμό. Δεν είναι απλή η ιδέα του να υπάρχει ένα κοινό εκπαιδευτικό σύστημα. Γλωσσικές δεξιότητες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ενδεχομένω, η πολυγλωσσία που φαίνεται να είναι το πρώτο και πιο εύκολο προϊόν του Erasmus Plus. Δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε το πιο εύκολο, το πιο αναγκαίο. Και τώρα προσπαθεί κανείς ε, να ε, επικοινωνήσει με τους ε, συνομιλίκους του από μια άλλη χώρα, σε οποιοδήποτε χώρα, προετοιμάζει τους ανθρώπους. Αυτή η πολυγλωσία είναι μία επιπλέον δεξιότητα. Δεν είναι όμως κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Η διγλωσία στην, ε, μεταξύ εκπαιδευτικών οργάνων, ε, ε, Ιδρυμάτων είναι ένα άλλο θέμα και νομίζω ότι θα πρέπει η ανακοίνωση να είναι τουλάχιστον σε δύο γλώσσες, η εκπαίδευση σε διάφορες γλώσσες είτε μιλάμε για τη Γερμανία, είτε μιλάμε για τη Ρουμανία, είτε μιλάμε για την ε, Λιθουανία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε μία μάχη. Νομίζω ότι απάντησα. Α, μάλιστα, μάλιστα. Οι εγγύησει για τα δάνεια, μάλιστα τα φοιτητικά δάνεια. Νομίζω ότι τα γεγονότα είναι πάρα πολύ εύλογα. Δόθηκαν αυτά τα δάνεια, τα φοιτητικά δάνεια σε 200.000 φοιτητέ. Ε, μόνο 300 τα χρησιμοποίησαν και αυτό για διάφορους λόγους. Καταλαβαίνω ότι σε ορισμένες σχόλες μέλη δεν ήταν κοινό, δεν είναι πολιτιστικά αποδεκτό ε, να παίρνουν οι φοιτητέ δάνεια. Και αυτό πρέπει να το ε, δεχτούμε. Σε άλλες χώρες ε, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ήταν τόσο πολύπλοκη, υπήρχαν τόσα διοικητικά μέτρα που ε, προτιμήθηκε η λύση του προσωπικού δανείου από την τράπεζα. Αυτό είναι κάτι που συναντάτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το πρόγραμμα Juncker είναι ένα από αυτά. Εάν δημιουργηθεί ένα τόσο μεγάλο διοικητικό, τόσο μεγάλος διοικητικός μηχανισμός και δεν σκεφτεί κανείς ε, τα κίνητρα, όλοι οι παίκτες, οι φοιτητέ ε, και οι μαθητές και άλλοι που θα μπορούσαν να δώσουν ε, πιστώσεις και εδώ βεβαίως το ρόλο το βασικό το παίζουν ε, οι αναπτυξιακές τράπεζες που είναι δημόσιες, όχι ιδιωτικές, θα ήταν μια λύση. Θα μπορούσαμε να τους προσεγγίσουμε προκειμένου να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση. Αλλά το θέμα παραμένει ανοιχτό και νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Για την ώρα ε, ε, αφήνουμε κατά, ε, ε, ε, κατά μέρος αυτό το μηχανισμό διευκόλυνση χορήγηση δανείων. Ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει δύο το λόγο. Κύριος Φραντς, καταρχάς. Σας ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι οι Ρωμά, παραδείγματος χάρη και άλλοι, ζουν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας και δεν έχουν πρόσβαση σχεδόν καθόλου στο Erasmus Plus, έχοντας ε, δε υπόψη και μία ακαδημαϊκά ε, επαγγέλματα. Θα ήταν σημαντικό να ε, έχουμε περισσότερους συμμετέχοντες, γιατί υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Η κοινωνική υποβάθμιση, κοινωνικό προβληματικό υπόβαθρο πρέπει να οριστεί, γιατί έχουμε το πρόβλημα ε, του ε, αντιτσιγκανισμού, αν μπορώ να το πω έτσι. Ε, και υπάρχει ένας πολύ σημαντικός διαχωρισμός ε, στη, στο εκπαιδευτικό σύστημα και θα μπορούσε αυτό ε, το που είπα αυτός ο αντι, αντι, ε, ε, αντισημιτισμός και τα λοιπά θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο το προσέχουμε ιδιαίτερα στη διδακταία ύλη για να το απαγορεύσουμε. Αν λάβουμε υπόψη τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη νομίζω θα δίναμε έτσι ένα πολύ καλό μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπίλτ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μαθαίνω στην εκθέση αυτή ότι χάρη στον χάρτη όπου αναφέρονται τα κατοικένα ιδρύματα βλέπουμε αύξηση της συμμετοχής ε, των ε, μειονεκτούντων ατόμων στο Εράσμους. Σίγουρα ε, οι ανισότητες τις βλέπουμε και στην κινητικότητα των ατόμων αλλά και στις σχολικές τους διαδρομές. Όμως αν το Εράσμους επέτρεπε στους ανθρώπους να ζήσουν μια εμπειρία εμπλουτισμού σίγουρα θα ήταν η ευκαιρία να εμβαθύνουν και στις ε, δεξιότητες. Τουλάχιστον μπορούμε να αναμένουμε από το Εράσμους ότι μπορεί να επιτρέψει στους ανθρώπους ε, να μάθουν καλά μια ξένη γλώσσα. Δυστυχώς δεν ισχύει πάντοτε κάτι τέτοιο όπως λέει η έκδοση. Η αξιολόγηση που έχει γίνει μας έχει δείξει ότι οι γλωσσικές δεξιότητες ε, δεν έχουν αλλάξει, μάλιστα έχουν μειωθεί. Γι' αυτό προσυπογράφω τη σύσταση της έκθεσης αυτής να ε, αποκαταστήσουμε την παραδοσιακή χρηματοδότηση για τη διδασκαλία στις αίθουσες και προτείνω να πάμε πιο μακριά, να καταστήσουμε υποχρεωτική την παρακολούθηση ενός μάθημα που να επιτρέπει ε, το να ε, διδαχτεί η γλώσσα, η επίσημη γλώσσα μιας χώρας υποδοχής. Ακόμη και αν ε, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι κάπως απογοητευτικά, αυτό ουσιαστικά θα συμβάλλει στο να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό αίσθημα των συμμετεχόντων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εσείς, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ειλικρινά, δεν έχω πολλά να προσθέσω, πέρα από το ότι συμφωνώ πλήρως με τις προτάσεις σας. Βεβαίως, η καταπολέμηση του ρατσισμού θα μπορούσε να είναι ένα επιπλέον στοιχείο της ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας, χρησιμοποιώντας ε, κάποια μέσα ή θέτοντας ε, προτεραιότητα, ε, σε προτεραιότητα κάποια προγράμματα όπου υπάρχουν τέτοιες ανάγκες. Θα μπορούσαμε εκεί να αντιμετωπίσουμε αυτά τα στοιχεία. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα ότι πρέπει να έχουμε μια ορθή οικονομική διαχείριση δεν μιλάμε για μια φούσκα, μιλάμε για το ότι δίνουμε χρήματα για να έχουμε ένα κοινωνικό αποτέλεσμα, η επίτευξη του οποίου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς ε, ευρω... σε ευρωπαϊκο... δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φυσικά η διδασκαλία στις αίθουσες, στην ελεγκτική ομάδα, όταν ε, μάθαμε τα στατιστικά στοιχεία, κάποιοι, όπως σωστά μας είπατε κυρία Μπίλτ, Κάποιοι φάνηκε να ε, έχουν επιδεινώσει τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Όμως, από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν δίνουν προσοχή στο γλωσσικό τμήμα του Erasmus Plus, απλώς συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο και συνεχίζουν ως έχει. Η διδασκαλία στην αίθουσα Απαιτεί οι άνθρωποι να έχουν φυσική παρουσία και τότε θα υπάρξουν και τα αποτελέσματα. Εκεί θα έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Και μάλιστα μπορείς και αντικειμενικά να ελέγξεις στη συνέχεια. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της δασκαλίας που χρηματοδοτείται από το Erasmus Plus, γιατί τα τεστ θα ε, τα ε, παρακολουθεί στη συνέχεια ένας ε, πραγματικός άνθρωπος με φυσική παρουσία. Στην επαγγελματική κατάρτιση, όπως σας ανέφερα και επιμένω, ε, οι μαθητές είναι πολύ καλή πηγή και ακόμη περισσότερο αν ε, δούμε τι συμβαίνει στην ανώτερη εκπαίδευση. Είδαμε σε κάποια κράτη-μέλη ότι ήδη υπήρξε ένα επίπεδο κορεσμού χρηματοδότησης των αιτήσεων. Έτσι λοιπόν, αν δεν διευρύνεις τη βάση, θα έχεις ε, προβλήματα ε, που να δαπανίσεις τους πρόσθετους πόρους. Εγώ πιστεύω όμως ότι χρειάζονται αυτοί οι πρόσθετοι πόροι και ότι θα δώσουν αυτή την προσθεμένη αξία. Θα εμπλέξουν δηλαδή και τους ανθρώπους που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα σε κάποιες δραστηριότητες ε, πολύ θετικές. Έτσι λοιπόν συμφωνούμε με αυτά που προτείνατε εμείς από την πλευρά του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt gerne noch Frau Eriksen von der Kommission das Wort geben. Frau Eriksen, bitte. Εσείς ε, ε, για δύο-τρία λεπτά θα πάρετε τώρα το λόγο. Thank you very much, Mr. President. Ich Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την πλευρά της Κομισιόν καλωσορίζουμε αυτή την ε, θετική έκθεση. Βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο έχει εντοπίσει πολλούς σημαντικούς ε, τομείς ε, όπου χρειάζεται βελτίωση και η Κομισιόν ε, συμφωνεί ότι μπορούμε να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες σε αυτούς τους συγκεκριμένου τομείς. Για το μελλοντικό πρόγραμμα θα κάνουμε προσπάθεια να προσπαθήσουμε ήδη να εφαρμόσουμε κάποιες από τις συστάσεις που έχετε θέσει επιτάπητος. Επίση, σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι πολλά από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έκθεση είναι παρόμοια με τη δική μα αξιολόγηση του προγράμματο. Είχαμε πολλέ διαβουλευσει και αξιολογήσει και είδαμε ότι υπάρχει ε, ουσιαστικά ένα μεγάλο συνδεσμός μεταξύ των δύο εγχειρημάτων και αυτό μα επιβεβαιώνει ότι ακολουθούμε τη σωστή οδό. Και όλα τα θετικά στοιχεία που τονίσατε, το brand name, ευρωπαϊκή προσταμενή αξία, η ενδυνάμωση του προγράμματο. Ε, ουσιαστικά ώστε να ξεπεραστεί η νομική του βάση. Όλα αυτά που τονίσατε επιβεβαιώνονται και στη δική μας έκθεση. Τα σημειώνουμε λοιπόν όλα αυτά. Κάποια παραδείγματα όπου βλέπουμε ήδη βελτιώσεις ε, και αναφέρατε κι εσείς κάποια, απλώς να επιβεβαιώσουμε και εμείς ότι πρόκειται για σημαντικές αλλαγές. Καταρχήν, τα όσα είπατε για το ε, να προωθήσουμε περισσότερο τους τομείς που έχουν ε, μικρότερη κρίσιμη μάζα, δηλαδή παραδείγματο χάρη να αυξήσουμε την κινητικότητα μεταξύ των ε, μαθητών στα σχολεία. Αυτό το έχουμε συμπεριλάβει στις μελλοντικέ μας προτάσεις. Επίσης, τα είπατε, για τις πτυχές ένταξης, στη δική μας πρόταση προσπαθήσουμε να το αντικατοπτρίσουμε αυτό με έμφαση, όχι τόσο στην έκθεση, αλλά το αναφέρεται αυτό τώρα, τη σημασία του να έχουμε πλήρη αναγνώριση και ε, έγκριση των περίοδων μάθησης που έχουν δαπανηθεί στο εξωτερικό. Αυτό ε, έχει να κάνει ε, με αυτό που βλέπουμε ότι αν δεν έχουμε αυτή την αυτόματη αναγνώριση, δεν θα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερα και ισχυρότερα προγράμματα. Εκτιμώ που και προφορικά. Επίσης, ε, κατανοώ την ε, κριτική απέναντι στα φτητικά δάνεια, το έχουμε αφαιρέσει από την πρόταση και επίσης ε, τονίσατε όλο το θέμα της δουλειάς απλούστευσης. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά να είναι πιο προσβάσιμο το πρόγραμμα, πιο φιλικό προς το χρήστη και να απλουστευτούν οι διαδικασίες της υποβολής εκθέσεων αλλά και των υποβολής αιτήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα τα σχόλιά σας για το πρόγραμμα. Ευχαριστώ την Κομισιόν. θα μπορούσε ίσως ε, η Κομισιόν ε, να πάρει μια-δυο μαθήματα από το Ελληνικό Συνέδριο για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η υποβολή αναφορών. Θέλετε να πείτε κάτι ακόμη? Ναι. Δεν έχω πολλά να πω. Αλλά στην προηγούμενη ζωή μου όταν ε, ήμουν δημόσιος υπάλληλος στη χώρα μου, είδα ότι αν εισάγεται κάποια διαδικασία επιβολής εκθέσεων, φυσικά μεγενθύνεται, μεγενθύνεται, μεγενθύνεται και χρησιμοποιούμε εκεί αυτή την ε, τεχνική ορολογία. Έτσι λοιπόν, εγώ θα συμβουλευά να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε αυτή την ορολογία, αυτή τη γλώσσα και να αφήσουμε ε, την υποβολή εκθέσεων που είναι μόνο σχετική. Και ίσως μία άλλη πρόταση που ήδη το φαντασιώνουμε, μερικές φορές είναι δυνατό να αλλάξουμε το βάρος της απόδειξης και να το μεταθέσουμε στους θεσμούς και να μην επιβαρύνουμε τους ίδιους τους φοιτητέ, να συμπληρώνουν πάρα πολλά έγγραφα που είναι στερεοτυπικά και τα ίδια ιδρύματα. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια ακόμη πρόταση όμως για τους δείκτες Πιστεύω ότι συνεχίζεται η συζήτηση. Ήδη είδα την έκθεση του κ. Σβέρ με τις προτάσεις για το πώς ε, θα βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν σε σχέση με τους δείκτες μέτρησης της επιτυχίας του προγράμματος. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Σας ε, εύχομαι έναν πολύ παραγωγικό τριμερή διάλογο με την Κομισιόν και το Συμβούλιο και φυσικά ανυπομονώ για τις μετέπειτα συζητήσεις που θα αφορούν τον κανονισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εμείς βάζουμε τα δυνατά μας για να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Σάτσιους και για την παρουσία σας και για την παρουσίαση της έκθεσης. Μπορείτε να παραμείνετε βέβαια για να ακούσετε και τον κύριο Σβέρ ο οποίος θα μας παρουσιάσει τώρα τις ε, δικές του προτάσεις, οποίες και στη συνέχεια θα συζητήσουμε, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Και τώρα πηγαίνουμε ευθύ αμέσως στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης, που είναι η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης για το νέο πρόγραμμα Εράσμους. Έτσι θα λέγεται από εδώ και πέρα. Το είπα πολλές φορές, ηγετής ο κύριος Βέρ και η προθεσμία κατάσταση τροπολογιών είναι στις 3 ε, το μεσημέρι, η 15 Νοεμβρίου, τα 13 Νοεμβρίου. Εσείς έχετε το λόγο κύριε Σβέρ τώρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή πρόεδρε, αγαπητή Σκιώδης, Αγαπητοί συνάδελφοι, φαντάζομαι ότι έχετε λάβει τις ε, τροπολογίες με τον ταϊτή ε, προσεχή κύκλο του Erasmus ε, Plus που τέσσερις μήνες πριν δημοσιοποίησε η Κομισιόν και είναι μια πολύ καλή αφετηρία. Έχουμε τη δομή με τους τρεις πυλώνες, δεν έχουμε εδώ κάποια διαφοροποίηση και αυτό είναι κάτι θετικό γιατί για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλουμε τέτοιους κραδασμούς σαν αυτούς ε, του 2014, ε, εξού και έμεινε άθικτη η βασική δομή του προγράμματος. Επίσης, ε, μπορώ να συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις τρεις νέες πρωτοβουλίες, δίκτυο με τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, Σκαβριγιού και το Κέντρο Αριστείας. Επίσης, θα πρέπει να εστιάσουμε και στις μικρές εταιρικές σχέσεις, ε, διευκόλυνση πολυγλωσσίας, ε, διευκόλυνση ανταλλαγής ε, μαθητών και προπονητών, αθλητών κτλ. Ε, όμως νομίζω ότι υπάρχουν βελτιώσεις που θα έπρεπε να είναι στη διαφάνεια, την ένταξη και την απλούστευση. Διαφάνεια πρώτα απ' όλα. Αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο προπολογισμό να είναι ε, ο ίδιος με αυτόν στον πρώτο κανονισμό και τριπλάσιος να είναι ο αριθμός ε, των ε, σπουδαστών που θα καλύπτεται. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να γίνει. Πρέπει όμως να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ αυτών που θα ε, είναι αντικείμενο της μακροχρόνιας κινητικότητας, αυτό κάποιο που δεν θα ε, μετακινούνται και κάποιοι θα συμμετέχουν σε βραχυπρόθεσμες ε, ανταλλαγές. Η ποιότητα πρέπει να προηγείται της ποσότητας. Εδώ και προτείνουμε κάποιους σαφείς ορισμούς. Το δεύτερο είναι η ένταξη. Το Erasmus Plus θα πρέπει να μπορεί να είναι προσβάσιμο από όλους τους κοινωνικού υποβάτου. Δεν είναι δεκτό μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν την οικονομική υποστήριξη των γονέων τους να μπορούν να ωφελούνται από τις μακροχρόνιες αυτές ανταλλαγές σπουδαστών. Εξού και προτείνω να συμπεριληφθούν διατάξεις που θα περιλαμβάνουν όλους τους σπουδαστές φοιτητές τουλάχιστον το 50% του κόστους της ανταλλαγής να καλύπτεται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Άλλοι μηχανισμοί, τα κράτη-μέλη θα καλύψουν το υπόλοιπο 50%. Τι μπορούμε να κάνουμε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα υποβάλουν αναφορά για τα προγράμματα και τα προβλήματα που ενδεχομένω έχουν αντιμετωπίσει. Η τρίτη αρχή είναι η απλούστευση. Τι προτείνω. Μία ενιαία θηρίδα γραμμική που μπορεί να χρησιμοποιείται και σε κινητές συσκευές, φορητές. Γιατί ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και πιστεύω ότι αν όποιο θέλει να υποβάλει μια αίτηση για να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγή κτλ., θα πρέπει με λίγα κλικ να μπορεί να τα καταφέρει. Η Κομισιόν επίση θεωρεί ότι οι αιτήσει ποιοτικέ θα πρέπει να χρηματοδοτούνται και από τα διευθυντικά ταμεία. Πώς θα γίνει αυτό. Πώ θα είναι επιλέξιμο ο ετών από, ένα, από τα διευθυντικά ταμεία ή τα επενδυτικά ταμεία. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει απευθείας η χρηματοδότηση να παρέχεται από τα διευθυντικά ταμεία απευθεια η χρηματοδοτηση να τροποποιηθεί ε, το project στο πλαίσιο του Εράσμού. Αν κάνουμε μια σύγκριση με τον κανονισμό, τον σημερινό και το μελλοντικό, θα δούμε τι είναι πιο σύντομη η νέα πρόταση. Δεν έχει, έχει μάλλον μεγαλύτερη ευελιξία η Κομισιόν. Σίγουρα μπορεί να ανταποκρίνεται και στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Δεν υπάρχει επίσης αναφορά στον κανονισμό για τα πόσα πόσα θα δαπανηθούν για αυτό το δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, το Discover You. Εντάξει, είμαστε στην αρχή, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω απαραίτητα. Καταλαβαίνω ότι θέλει μεγαλύτερη ευελιξία η Κομισιόν, αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο ως Κοινοβούλιο και να συμμετέχουμε και στην εκδοτήση προγράμματος εργασίας που θα καλύψει και όλες τις λεπτομέρειες που δεν αναφέρονται στον κανονισμό. Θέλουμε δηλαδή περισσότερες καταξιοδότηση πράξη και λιγότερες ε, εκτελεστικέ. Σε ό,τι διαφορά τον προπολογισμό, τον Ιούνιο είχα πει ότι αν θέλουμε τριπλασιασμό προπολογισμού θα έχουμε περισσότερους φοιτητές ταυτόχρονα. Δύο πυλώνε έχει το πρόγραμμα, δύο σκέλη. Θα μπορούν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγή φοιτητέ. πιο εύποροι και οι πιο ε, λιγότερο εύποροι σε εικονικά προγράμματα. Καλό είναι και αυτό, αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν είναι υποκατάστατο ενός προγράμματος ανταλλαγής. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των κοντιλίων, δεν ασχοληθήκατε ιδιαίτερα με την πρόταση της Κομισιόν, γιατί ξέρω ότι όλοι θέλουν περισσότερα χρήματα, όμως δεν πρέπει να πάρουμε χρήματα από τις ανταλλαγές παιδιών και να πάνε αυτά τα χρήματα σε ενήλικους, στον αθλητισμό ή στην νεολαία. Θα πρέπει να είναι αύξηση, η αύξηση του προπολογισμού τεράσμου συνολική. Σε ό,τι δε αφορά την ονομασία του προγράμματος, νομίζω δεν πρέπει να ειναι αυξηση η αυξηση του προϋπολογισμού τερασμου συνολικη σε οτι δε αφορα την ονομασια του προγραμματος νομιζω δεν πρεπει να αλλαξει Στι επόμενε μεσονομικές προοπτικέ, γιατί πλέον θεωρείται το σε ένα πολύ υψηλό πρόγραμμα ανταλλαγή και εν ώψη των ευρωεκλογών. Θα ήταν καλό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και σε ό,τι αφορά τη δική μου την έκθεση. Δεν εξαρτάται όμως όλα από μένα και τους ε, ειδικού που με βοηθούν. Θα πρότεινα λοιπόν, αν αυτό είναι δυνατό, να κατατεθούν στο δυνατόν περισσότερες τροπολογίες από κοινού με τις άλλες πολιτικές ομάδες και βασίζομαι στη δική σας υποστήριξη. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να μου καταθέσετε επικοδομητικές τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεσή μου, κάθε της λέξη βασίζεται σε μια συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία είναι βελτίωση του προγράμματος. Μπορείτε να ήρθατε σε επαφή με τον Νταρένου Νεβίλ, ε, τον Ντάρεν Νεβίλ ή τον Μάρκους Προύτς, οι οποίοι και εγώ βέβαια είμαστε στη διάθεσή σας να σας απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα περνάμε στους σκιώδεις εισηγητές. Όσοι είναι εδώ ή εκπροσωπούνται. Όπως παραδείγματος χάρη η κυρία Λιμπάτσκα που εκπροσωπείται από την κυρία Κώστα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα διαβάσω την παρέμβαση της συναδέλφου Ριμπάσκα ως κοιόδης συγγητρίας. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την πληρέστατη έκθεση. Χαιρόμαστε που πολλά από τα θέματα που συζητήσαμε και ε, συμπεριλήφθησαν σε αυτό το σχέδιο έξεση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα σημεία. Η ομάδα μα με χαρά θα παρουσίασε περαιτέρω προτάσει για να ισχύσει μερικέ ε, πτυχέ του προγράμματο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. ό,τι αφορά τον προπολογισμό, συμφωνούμε ω προ την ανάγκη τριπλασιασμού του, όπω προβλέπετε στο ε, ψήφισμά μα πλαίσια του νέου ΜΜΕΦ Είμαστε υπέρ μια γραμμική αύξηση των κονδυλίων του προπολογισμού. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το πρόγραμμα να οδηγεί στην ένταξη. Η κοινωνική ένταξη είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τα άτομα που έχουν λιγότερε ευκαιρίε συμμετοχή. Προκειμένου το πρόγραμμα να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να λάβει υπόψη του μία επιπλέον υποστήριξη για αυτού που είναι σε μειονεκτούσα θέση, μεταξύ των οποίων, αλλά όχι κατά αποκλειστικό, ε, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, το υπόβαθρο, οι γεωγραφικές, πολιτιστικές, ε, ε, τα γεωγραφικά στοιχεία θα πρέπει βεβαίως να λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία, μέτρα για τη συμμετοχή ε, τα μέτρα για τη συμμετοχή θα ποικίλουν για ορισμένους, θα πρόκειται για οικονομική βοήθεια. Για άλλους μια καλύτερη μέρωση για το πρόγραμμα. Παρά όλα αυτά θα πρέπει η προσέγγιση να είναι ευρεία και ε, να υπάρχει μια πλήρη στρατηγική προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν αυτές οι ομάδες. Όλα αυτά θα πρέπει να ορίζονται σωστά στο πρόγραμμα. Παράλληλα, όπως είπε ο εισηγητής, χρειαζόμαστε τους κατάλληλους δείκτες για να μετρήσουμε την επίπτωση των δράσεων που προτείνονται σε Α, για τα δικά μου τα μέτρα διαβάζω πολύ αργά. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου στι ε, στρατηγικές ένταξει που προτείνονται από τον εισηγητή. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική σε επίπεδο ευρωπαϊκό, προκειμένου να υπάρξουν κοινά πρότυπα σε αυτό το επίπεδο που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν περαιτέρω σε επίπεδο εθνικό και τοπικό και να εφαρμοστούν από τους τοπικούς φορείς. Εκτός από αυτό, χρειαζόμαστε διευκρινήσεις ως προς τις νέες πρωτοβουλίες και τον προϋπολογισμό τους. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στο Discover You και στο ε, European Universities Network. Σε ό,τι αφορά τις συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων Horizon και Creative Europe, αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε επίπεδο προγραμματισμού και εφαρμογής. Σε επίπεδο προγραμματισμού χρειαζόμαστε μία πολιτική, σφαιρική συνεπή στρατηγική σε όλα τα σχετικά προγράμματα, καθώς και απολοποιημένες διαδικασίες για τους δικαιούχους σε επίπεδο εφαρμογής. Τι να κάνω σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη ε, αξία σε επίπεδο ευρωπαϊκό του προγράμματος, το Erasmus Plus είναι το έχει την καλύτερη προστιθέμενη αξία, αλλά θα πρέπει να αφήσει περιθώριο για τι καινοτομίε. Σε ό,τι αφορά τι προτεραιότητε του ετησίου προγράμματο, θα πρέπει να διατηρηθεί η συνέχεια και η ευελιξία. Γι' αυτό συμφωνούμε με τι κατεξουσιοδότηση πράξη. Τέλος, υποστηρίζουμε την εφαρμογή κανόνων σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκμάθηση ξένων γλωσσών, η ICAR κτλ ιδιαίτερη, να αναφέρουμε σε ορισμένα από τα βασικά σημεία, ε, διαρκής μάθηση, αυτό θα πρέπει να σα απασχολήσει ιδιαίτερα. Διατομεακή συνεργασία, μεγαλύτερο διάλογο με τα κοινωνικά, τους κοινωνικούς φορείς, ε, ε, είναι ενδιαφέρουσα η κινητικότητα του προσωπικού στα νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθμούς και ίση ανταμοιβή ε, ε, ε, για τους καθηγητές, τους ερευνητές και τους δασκάλους που ασχολούνται με τα ίδια προγράμματα. Τέλος, αυτό που υπογραμμίστηκε ήδη, όλα τα έγγραφα θα πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις επίσημες γλώσσες για τους δικαιούχους. Θα υποβληθούν προτάσεις και σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μια καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι πάντοτε δύσκολο να ε, διαβάζει κάποιο ένα κείμενο που δεν το έχει γράψει ο ίδιος. Ε, να λίγο πιο αυστήρη και συγγνώμη. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περίμενα να ακούσω την παρέμβαση του Ρόπου. Καταρχάς ήθελα να συγχαρώ για την έκθεση η οποία με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο σαν ομάδες ε, Η ε, ε, ΣΥΑΡ θα, υποβα... θα συμβάλλουμε και εμείς. Εμείς μιλάμε για τριπλασιασμό, όχι για διπλασιασμό. Γιατί, Γιατί θεωρούμε ότι σε τόσο δύσκολες εποχές για την πολιτική, σε μία εποχή που η πολιτική θα πρέπει να έχει ένα μακρόπνο όραμα, υπάρχει ανάγκη να γίνει μία μεγάλη επένδυση τα επόμενα 7 χρόνια. Θα έλεγα τα επόμενα 8 χρόνια. Θα ήθελα να αναφερθώ στο 14, 20, 21, 27 γιατί η θέση της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τους νέους είναι στρατηγική. Ε, είναι πολύ δύσκολο να προφέρει κανείς αυτή τη λέξη πολλά χρόνια μετά την υποδόμηση της ε, Ευρώπης. Θα καταλάβατε, αφού μιλάω Ιταλικά, ότι είμαι Ιταλός. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια έρχομαι σε επαφή με 28 χώρες και βλέπω ότι δεν με βρίσκει πάντα σύμφωνο η γενικότερη στρατηγική. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι το Εράσμους είναι ένα εργαλείο. Καταλαβαίνω αυτούς που λένε ας κάνουμε περικοπές από τη βιομηχανία, από την ε, γεωργία. Ε, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι και το Εράσμους Αναρωτιέμαι λοιπόν αν δηλαδή, είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή για να γίνουν επενδύσεις. Το 2017 είναι η στιγμή που διασχίζουμε την έρημο. Όπως σας είπα, συμφωνώ με την έκθεση. Θα ήθελα να πω ότι όταν ζητάμε έναν τριπλασιασμό της δαπάνης, υπάρχει ένας πολιτικός λόγος θα συνεργαστούμε με την, ε, τον ε, εισηγητή και με όλους προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στρατηγικός στόχος για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Δεν ε, είμαι η σκάδος της Βράσινης. είναι η κυρία Evans, αλλά δεν μπορεί να είναι εδώ. Θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια. Αυτό το πρόγραμμα, όπως ε, ακούσατε και το ξέρουμε εδώ και τι, είναι ένα πρόγραμμα ναρβαχίδα, είναι ένα πρόγραμμα επιτυχές και ε, για μένα αφορά την ενδυνάμωση διάφορων ανθρώπων, των μαθητών, των φοιτητών, ε, των μειονεκτούντων ανθρώπων, ακόμη και των παιδιών στα σχολεία, των νέων και των ενηλίκων. Και τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ε, σκεπτικισμό απέναντι στη σελίδα. Αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ καλό γιατί μα δείχνει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια πηγαίνουν κατευθείαν σε άτομα, σε ανθρώπου και με τι ε, ερχόμενε εκλογέ και με τη συζήτηση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό είναι ένα σημαντικό επιχείρημα γιατί αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα και μπορούμε να δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι για αυτού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε «Α, ξέρουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας» και νομίζω ότι με αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να δείξουμε ότι κάνουμε πολλά για αυτούς και ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερα. Επομένως, είναι σαφές ότι πρέπει να αυξήσουμε τον προπολογισμό, συμφωνώ απόλυτα, πλούστευση και όπως γνωρίζουμε πάντοτε αυτό ε, είναι σωστό γιατί εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το πρόγραμμα. Σε σχέση με το θέμα γιατί αν θα πρέπει να είναι μονοψηφιακό εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Γιατί εάν και εφόσον ε, θέλουμε να απευθυνθούμε σε μειονεκτούντες νέους ή με λιγότερες ευκαιρίες και δυνατότητες, νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε και ε, αναλογικές αιτήσει. Ο τίτλος για μένα είναι εντάξει, όπως είπατε, Ξέρουμε ότι είναι ένα εμπορικό σήμα, δεν πρέπει να αλλάξει ένα εμπορικό σήμα και ένα άλογο που κερδίζει, πάντοτε πρέπει να το διαφυλάσει. Και σύμφωνα με όσο υπόθηκαν, μεγαλύτερη ευελιξία, αυτό είναι καλό τρόπο να απευθυνθούμε σε νέου, σε μειονεκτική θέση και να έχουμε μια πολιτική συζήτηση τώρα με το πολιτέ πλαίσιο και τι μελλοντικέ εκλογέ. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα ως Επιτροπή Πολιτισμού, γιατί έχουμε ισχυρά επιχειρήματα που μας υποστηρίζουν. Η κυρία Μπίλτ. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Προτείνεται τριπλασιασμό του προπολογισμού ε, ενώ ο στόχος της Κομισιόν είναι να τριπλασιάσει τον αριθμό των ε, συμμετεχόντων. Να δούμε αντίστροφα, ε, είμαστε λογικοί. Ε, το πρόγραμμα Εράσμους λειτουργεί καλά, ας μην μειώσουμε την ποιότητα επειδή θέλουμε κάτι γιγάντιο. Ο διπλασιασμό του προπολογισμού που προτείνεται από την Κομισιόν είναι ήδη κάτι έκτακτο. τώρα, σε ό,τι αφορά το Discovery U, ε, δεν υπάρχει καμφιβολία ότι οι νέοι που μπορούν να είναι κάτι επίστευτο και ακριβώ αυτό με κάνει δύσπιστη. Είμαστε ένα έτος πριν τι εκλογές, η Κομισιόν αποφασίζει να κάνει εξαιρετικά δώρα στου 18 χρονου δηλαδή σε αυτού που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και ε, ανήκουν στην ηλική ομάδα που ψηφίζει λιγότερο. Συνήθω τα ραδιόφωνα δίνουν δωρεάν ταξίδια στου ακροατέ και σε ένα εμπορικό πλαίσιο. Ποιο είναι εδώ ο σκοπό τη Κομισιόν. Ε, επίσης, ε, ε Βλέπουμε ότι η Κομισιόν δεν ε, αιτιολογεί την ύπαρξη του Discovery U, απλώς ε, λέει ότι δίνει 7 εκατομμύρια ευρώ στο ε, προπολογισμό του Εράσμου. Έχετε δίκιο να απαιτείτε περισσότερη ευκρίνεια για τη λειτουργία του. Ας ζητήσουμε λοιπόν από την Κομισιόν να αποδώσει και τους λογαριασμούς, να λογοδοτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει και το θέμα της συνέργειας ε, ή των συνεργειών με άλλα προγράμματα. Και θα ήθελα και είχα μιλήσει με τους ε, συντονιστές των Επιτρόπων Αύρεσιτς και την να μου πούν ε, πώς γίνεται αυτό και πώς μπορεί να υπάρξει συνέργεια. Γιατί υπάρχουν και διαφορετικά ε, ε, διαφορετικές τα νομή κονδυλίων. Υπάρχουν και από τα κράτη-μέλη κάποια προγράμματα και οι αποφάσεις λαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο. Πήραμε κάποιες αποφάσεις τελευταία των συντονιστών να καλέσουμε σε συνάντηση των συντονιστών ε, τους επιτρόπους ώστε να μας ε, πει τι ακριβώς θα γίνει ε, σε επίπεδο κατών μελών. Καλές οι συνέργειες, στην πράξη όμως πώς λειτουργεί. Γιατί τελικά είναι μια λευκό εξοδότηση για την ε, Κομισιόν που μπορεί να αλλάζει άνετα και να πηγαίνει τα χρήματα από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες εξηγήσει για το πώς αυτά θα λειτουργήσουν ουσιαστικά στην πράξη. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε τον Επιτρόπο να μας τα εξηγήσει από κοντά. Α, ναι. Μια παρατήρηση προσωπικά, μιλάω τώρα όχι ως πρόεδρος, παραδέχομαι ότι Κάπως δυσκολεύομαι με το Discovery you. Ούτε έχω καταλάβει από το κείμενο περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Υπάρχει έννοια, αλλά δεν περιγράφεται κάπου και καλό θα ήταν να το διατυπώσουμε κάπως καλύτερα και πιο συγκεκριμένα. Ότι έχει να κάνει με τη μαθησιακή κινητικότητα κινητικότητα αλλά και μάθησιακή, γιατί η μάθηση είναι αυτό που πρέπει να είναι στο επίκεντρο ενός προγράμματος όπως το Εράσμους και νομίζω πρέπει να το τονίσουμε λίγο πιο πολύ. Και επίσης καλό είναι να προσπαθήσουμε να συγκεκριμενοποιούμε λίγο τα πράγματα και πράγματι να μην ε, προσφέρουμε ένα δωράκι σε κάποιον ή να πάει τρεις εβδομάδες σε μια ευρωπαϊκή πόλη γιατί τελικά αυτό δεν είναι και αρκετό. Ο κύριος Βέντα θέλει τώρα το λόγο. Θα συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τα σχόλια για το Εράσμο. Θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή μου σε ένα σημείο. Δεν συμφωνώ με την τροπολογία 26 σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Αν στόχος του προγράμματος αθλητισμού είναι η υποστήριξη του αθλητισμού, όπως αναφέρεται στο εκτιμώντας 13, έχει νόημα να παρέμβουμε σε αυτό το επίπεδο. Το δεύτερο σχόλιο Στο, στην τροπολογία 28 μιλάμε για την κινητικότητα και στον τομέα του αθλητισμού. Αυτό όμως θα πρέπει να το προσδιορίσουμε. Γιατί μερικέ φορές αναφερόμαστε στα άτομα που έρχονται από μία επιτροπή, την Ολυμπιακή Επιτροπή, για παράδειγμα. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να περιλάβουμε έναν ορισμό και για αυτούς τους ανθρώπους. Ενδεχομένως από το Συμβούλιο θα, θα πρέπει να, γίνει, να δοθεί ένας ε, σαφής ορισμός τι, τι εννοούμε, αν μιλάμε για άτομα που αμείβονται, αν μιλάμε για άτομα που εργάζονται πεθελοντικά. όταν φεύγουν από τη χώρα τους υπάρχει μία σύμβαση. Τώρα μία επιπλέον ερώτηση για τις τρίτες χώρες. Άρθρο 16 17. Μέχρι ποιο σημείο φτάνουμε σε ό,τι αφορά τον ορισμό των εταίρων από τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Κυρία Έριξ άλλη μια φορά εσείς το λόγο από την Κομισιόν. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο και μεγάλη χαρά άκουσα τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που έγιναν. Από τη δική μας πλευρά συμφωνούμε απόλυτα, απόλυτα ότι το Εράσμους είναι πραγματικά η ναυαρχίδα των πρωτοβουλειών και νομίζω ότι απευθύνεται άμεσα στους νέους της Ευρώπης. Από πλευράς Επιτροπής ε, σαφώς μας βρίσκει σύμφωνο το σχέδιο έκθεσης και πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις προτάσεις Επιτροπής. Βεβαίως και εμείς ελπίζουμε για μια αύξηση του προπολογισμού γιατί όπως είπατε και εσείς, προηγείται η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Χρειάζεται λοιπόν επαρκής ε, ε, προϋπολογισμός ε, για να καλυφθούν οι διάφοροι τομείς του προγράμματος και να αποκτήσουν πρόσβαση όλο και περισσότερα άτομα. Σε ό,τι αφορά άλλα σημεία, θα ήθελα να πω με ποια συμφωνούμε. Καταρχάς, το βουλευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να οδηγεί στην ένταξη, να προωθεί την ένταξη. Αυτό το έχουμε και στη δική μας πρόταση και αναφέρεται και στο σχέδιο έκθεσης ε, για μας η ένταξη αφορά, έχει πολλές διαστάσεις. Ε, θα πρέπει να δούμε το σύστημα των υποτροφιών, θα πρέπει ενδεχομένως να υπάρχει μια στρατηγική, όπως είπε από τους ε, ομιλητή, ομιλητής, καλύτερη προσβασιμότητα για όλους. Θα ήθελα όμως να έχω την βεβαιότητα ότι σε ό,τι αφορά τον τύπο και την κινητικότητα ε, να έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι τα βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Μιλώντας για συνέργειες, το είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι προσπαθήσαμε να δουλέψουμε προετοιμάζοντας τους διάφορους κανονισμούς ε, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό ESF, ΣΥΝ και Εράσμους, είδαμε άλλες παρόμοιες διατάξεις να σας παραθέσω ένα παράδειγμα του τι εννοώ πρακτικά. Θέλουμε δηλαδή να υπάρχουν επιπρόσθετα ωφέλη, να μπορούμε να προσθέτουμε ε, ε, ωφέλη για συγκεκριμένη ομάδα, ε, για συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό γίνεται στην Πολωνία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται πιο συχνά. Επίσης αναφερθήκατε στο θέμα της απλοποίησης και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να αναφέρω αυτό που αναφέρεται στην έκθεση. Αναφερθήκατε στην ενιαία θηρίδα. Υπάρχει ένα, το Erasmus Plus και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Κάρτα των φοιτητών, που αυτό πραγματικά δίνει μεγάλο δυναμισμό στο πρόγραμμα, προκειμένου να γίνει πιο φιλικό πιο προς το χρήστη. Υπάρχουν ορισμένα σημεία της έκθεσης με τα οποία δεν συμφωνούμε απόλυτα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω δύο λόγια και για το Discovery U. Σε ό,τι αφορά την πρόταση και το όνομα, η δική μας λογική ήταν ότι ήταν θετικό το να υπάρχει ε, κινητικότητα στο Εράσμους. Μετά από 7 χρόνια Εράσμους ε, με θεωρήσαμε ότι το πρόγραμμα ήταν ε, πλέον όριμο και να εγκαταλείψει με την προοπτική του 2027 το πλάσα. Δεύτερον, θα πρέπει επίσης να πω ότι μας προβληματίζει λίγο στο σχέδιο ε, έκθεσης η αναφορά σε κατεξουσιοδότηση πράξης. Κατά την άποψή μας έτσι μεταφράζονται οι νομικές διατάξεις σε ε, εφαρμοστικές διατάξεις, εφαρμοστική πράξη δηλαδή. Η ε, κατεξουσιοδότηση στην ουσία συμπληρώνει την νομοθεσία. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι και νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να παραμείνει εφαρμοστική πράξη. Τελευταίο σημείο, ελπίζω να μου δώσετε τη δυνατότητα να έχω λίγο περισσότερο χρόνο για να αρθετώ στο Discovery EU, σε αυτή την πρωτοβουλία, βεβαίω θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα να απλώ ότι λάβαμε, λαμβάνουμε υπόψη μας το αίτημα που ακούστηκε σε αυτή την αίθουσα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό που εφαρμόζουμε τώρα με αυτό που θα κάνουμε με αυτή την πρωτοβουλία όταν την εντάξουμε στο μελλοντικό πρόγραμμα Εράσμους. Οτιδήποτε στο μελλοντικό πρόγραμμα Εράσμους θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους και να έχει μία έντονη μαθησιακή διάσταση. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ότι ε, έχει εφαρμοστεί πιλωτικά σήμερα με αυτό που θα γίνει στο μέλλον. Η προπαρασκευαστική δράση θα μας βοηθήσει προσπαθήσει να σχεδιάσουμε τις μελλοντικέ πρωτοβουλίες. Και θα πρέπει να πω ότι 50.000 ε, νέοι ταξίδεψαν και έδωσαν, ε, οι απόψεις τους ήταν θετικές. Θα ήθελα να τονίσω ε, το ότι ο τρίτα από τους συμμετασχόντες είπαν ότι δεν θα είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη δίχως αυτό το πρόγραμμα. Αυτό μας λέει κάτι για τον χαρακτήρα του προγράμματος που οδηγεί στην ένταξη. Το 60% λένε ότι βελτίωσαν τις γλωσσικές τους γνώσεις. Είναι ε, ε, πολλοί, είπαν ότι έμαθαν πολλά για την πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη, μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με άλλους νέους ανθρώπους και μπόρεσαν να, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιλύσουν προβλήματα. Νομίζω μέχρι στιγμής ε, οι γνώμες που ακούστηκαν ήταν θετικές, βεβαίως ε, είναι περιορισμένος ο αριθμός αυτών που απάντησαν. Ε, στο το Νοεμβρίου θα έχουμε 12.000 επιπλέον συμμετέχοντες. Αυτό είναι ένα άτυπο μέρος του προγράμματος, δεν το είχαμε στο παρελθόν και είναι σημαντικό ότι αποτελεί ένα μια δράση που προωθεί άλλες ε, δραστηριότητες. Ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να λάβουμε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Τελειώνοντας, ε, θα ήθελα να πω ότι σας καλούμε να συνεργαστούμε μαζί αλλά και με άλλους ενδιαφερόμενους, με το Συμβούλιο για παράδειγμα, προκειμένου να προωθήσουμε την πρωτοβουλία αυτή με έναν ευρηματικό και δημιουργικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν θα πω τίποτα για το τέλος, αλλά θα πω κάτι για τις κατεξοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις. Είναι πραγματικά βασικό το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι στο Κοινοβούλιο Πραγματικά οι επιτροπές ε, είμαστε σύμφωνες. Εντάξει, να αφήσουμε κάποια περιθώρια ευελιξία σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή των προγραμμάτων στην Κομισιόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα επιτρέψουμε ε, σε κάθε πρόγραμμα εργασίας να αποφασίζονται με εκτελεστικές δράσεις για τις πολιτικές προτεραιότητες και έτσι να εγκρίνονται και πολιτικές προτεραιότητες. Εσείς δώσατε ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα που είναι το Discovery ναι, πράγματι πρέπει να αναπτυχθεί. Εντάξει. Αυτό θα γίνεται μέσα από τα αιτήσια προγράμματα εργασίας. Το Συμβούλιο όμως ε, και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι αυτά τα οποία θα θέτουν τις πολιτικές προτεραιότητες είτε μέσω ενός νομοθετικού κειμένου, το οποίο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, είτε μέσω μιας κατεξοδότησης πράξης που τελικά τουλάχιστον θα μπορούμε εμείς να πούμε όχι δεν το θέλουμε έτσι να γίνει αλλά όχι πλέον ε, να εφαρμόζονται πράγματα τα οποία εμείς ε, δεν τα έχουμε ορίσει ε, ως πολιτικές προτεραιότητες. Είναι κάτι που πάει πολύ πιο μακριά. Αν θέλετε ευελιξία, τότε θα σας πούμε κι εμείς ναι, εντάξει, συμφωνούμε, όμως με κατεξοδότηση πράξης. Αν θέλετε μόνο εκτελεστικές πράξεις, τότε εμείς θα γράψουμε τόσο αυστηρά ε, τις διατάξεις που δεν θα σας αφήνουμε κανένα περιθώριο ελιγμών. Και εμείς μαζί με το Συμβούλιο θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα θέτουμε τις πολιτικές προτεραιότητες. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική αντιπαράθεση αυτή μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να το περιορίσουμε στα τεχνικά ζητήματα. Δεν είναι τεχνική εφαρμογή αμυγός το θέμα. Δεν θέλουμε καμία παρέμβαση στις κατευθυντήριες γραμμές ή στο πώς ε, θα κατανέμονται και θα δαπανούν τα, τα κονδύλια. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το πώς θα πάνε τα πράγματα, ε, τις λεπτομέρειες. Αυτά κάντε τα με τελεστικές πράξεις αν θέλετε. Όμως όταν μιλάμε για ε, τις ε, πολιτικές προτεραιότητες μέσα από αιτήσια πρόγραμματα τότε θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να έχει και μια λεξούλα εδώ, θα πρέπει να έχει ένα λόγο το κοινοβούλιο. Το ξέρετε και εσείς κυρία Έριξεν, δεν αφορά μόνο τη δική μας επιτροπή, αλλά και πολλές άλλες ε, επιτροπές που το έχουν πει ξεκάθαρα, πρέπει να το ξαναπούμε ξεκάθαρα και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε σκληρά. Παναλαμβάνω, όταν μιλάμε για καθορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων, εμείς και το Συμβούλιο είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να έχουμε την ευθύνη γι' αυτό. Ε, ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σβέρ. Ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Πιστεύω ότι δεν ε, υπάρχουν πολλά προγράμματα της Ένωσης που χαίρουν ε, τέτοιο βαθμό συνένεσης όπως το Erasmus+. Κάποιες ιδέες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Επίσης, ε, η έννοια της ισότητας ως προς τις πληρωμές. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό όταν θα ολοκληρώσουμε την έκθεση. Τώρα, σε αυτό που ε, πρότεινε ο συνάδελφος ε, για την ε, διαγραφή του ορισμού της τρίτης χώρας. Ο πρώτος ε, ήταν αρκετά ευρύς και κατανοητό. δεν χρειαζόταν να έχουμε διορισμούς. Τώρα, σε σχέση με τη διαγραφή της τροπολογίας, που διαγράφει τον όρο grassroots sports, αυτό το έχουμε συμπεριλάβει ξανά στην έκθεση, αλλά χρειαζόμαστε μια τροπολογία. Τώρα ορίζεται μόνο στο πρώτο τμήμα, αλλά στη μέση της έκθεσης ουσιαστικά δεν μιλάμε για τον αθλητισμό σε επίπεδο βάσης, grassroots sports. Ίσως ε, θα έπρεπε να μου δώσετε μια τροπολογία ε, και στη συνέχεια μπορώ εγώ να αποσύρω τη δική μου. Εγώ συμφωνώ όμως επί μήπως ε, να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με την αξιολόγηση του Discovery U. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν πιστεύω ότι η τυπική εκπαίδευση είναι το πιο σημαντικό τμήμα. Και η άτυπη μάθηση είναι επίσης σημαντική. Οι νέοι όταν ταξιδεύουν στα πλαίσια του προγράμματος ε, κερδίζουν ε, κάποιες ε, δεξιότητες και γλωσσικές δεξιότητες. Πιστεύω ότι και η άτυπη μάθηση αλλά και μη τυπική μάθηση θα πρέπει να εκτιμηθούν εντός του πιλωτικού προγράμματος που θα τεθεί σε εφαρμογή με την πρωτοβουλία Discovery You. Επίσης ευχαριστώ την Κομισιόν που μας ε, παρουσίασε αυτά τα πρώτα επιχειρήματα. Νομίζω ότι θα ακολουθήσει μια καλή πορεία αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι μου δώσατε μια ισχυρή εντολή προκειμένου να μπορέσω να απαγιώσω τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Ίσως ε, θα ε, μπορέσουμε να έχουμε και διαπραγματεύσει εντό αυτής της θητείας. Σα ευχαριστώ πολύ. 22 Νοεμβρίου, 10 το πρωί. Όχι, τι λέω, 13 Νοεμβρίου, 3 το μεσημέρι. Αυτή είναι η προθέσμια για την κατάσταση των τροπολογιών. Κύριε Σφέρ, εύχομαι και σε εσά και στους και κάθε επιτυχία. Και είμαι βέβαια ότι θα κολλήσουμε κάπου, ε, αλλά ε, επί των βασικών είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Ήμουν την Παρασκευή σε μια εκδήλωση με 300 άτομα που γύρισαν από την Ευρωπαϊκή Θελοντική Υπηρεσία, όχι από το Σώμα Εθελοντών, από την την, το Σώμα από την Εθελοντική Υπηρεσία και ήταν πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με αυτά τα οποία έκαναν και μας έλεγαν συνεχίστε το, ενισχύστε το, βάλτε, το, βάλτε περισσότερα κονδύλια σε αυτό το πρόγραμμα μέσω του Erasmus+. Τουλάχιστον βλέπουμε να γίνονται κάποια πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοδομητική συζήτηση. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστεί και τους διερμηνείς ε, για την υποστήριξη η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και εμείς. Ξέχασα κανένα λέει Πρόεδρος, όχι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στην επόμενη συνεδρίασή μας που είναι στις 8 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.